σας και για την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας. Και χαίρομαι που είμαι η πρώτη επίτροπος που ε, συνεργάζεται μαζί σας υπό τη νέα σας αυτή ιδιότητα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα συγχαρητήρια που εκφράσατε. Ευχαριστώ άλλωστε και όλες και όλους που με συνεχάρισαν. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένα είδος κυβωτός του ΝΟΕ, μια κοινότητα αλληλεγγύης, στην οποία αναχωρούν πολλοί. Έξι ψηφίσματα ακολουθούν την συζήτηση αυτή, έχουν κατατεθεί για το θέμα. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτή. Αύριο θα γίνει η σχετική ψηφοφορία. Το τελευταίο θέμα στην απόψινή ημερήσια διάταξη και απευθύνω χαιρετισμό σε όλες και όλους που εξακολουθούν και παραμένουν εδώ απόψε. Έχουμε προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών. Θα παρακαλέσω πρώτα τον κύριο Μπελινγκουέρ να κάνει τη σχετική εισαγωγή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η προφορική ερώτηση και το σχετικό ψήφισμα προέκυψε γιατί θέλαμε να επισημάνουμε ότι στο σχέδιο δράσης της Στοκχόλμης είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ε, μια δικαστική ευρωπαϊκή κατάρτιση η οποία θα είναι διαδεδομένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα εν ώψη και τη ανακοίνωση τη οποία θα πρέπει να μα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μελλοντικά πιλωτικά προγράμματα, όπω μα είπε, να διευκρινίσουμε κάποιες έννοιες. Καταρχάς, θα πρέπει να ξεκινήσουν σύντομα οι διαβουλεύσεις ε, και οι διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όταν θα αρχίσει να σκιαγραφείται αυτή η ιδέα των ε, μελλοντικών ε, προγραμμάτων, να έχει γίνει εγκαίρος και να υπάρχει και δική μας συμμετοχή, να μην είμαστε οι τελευταίοι τροχοί της αμάξης. θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι ο εθνικός δικαστής, ο συνήγορος ε, κράτη-μέλη είναι σημαντική πτυχή στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, διότι λαμβάνοντας υπόψη και το εθνικό δίκαιο στα ευρωπαϊκά θύματα, δίνονται οι προϋποθέσεις για να επιλύονται οι διαφορές και να ρυθμίζεται η καθημερινή ζωή των πολιτών και έτσι να θεμελιωθεί η ευρωπαϊκή υπηκότητα, μια ευρωπαϊκή ταυτότητα για όλους όσους διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορούν να δουν οι δύο όμαση τα πλεονεκτήματα που προεκύπτουν για την, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα δικαιώματα των ανθρώπων και για το δίκαιο των κρατών μελών, κυρίως και για το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρχουν όλα αυτά τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από την επίλυση των προβλημάτων τα οποία εάν δεν υπήρχε το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν θα επιλύονταν. Θα θέλαμε μετά από όλα αυτά να ανατρέψουμε την όλη τοποθέτηση. Δεν θα θέλαμε όλα αυτά τα προγράμματα να είναι ε, στο στυλ του Εράσμους, διότι οι δικαστικοί που θα συμμετέχουν σε αντίστοιχα προγράμματα με αυτά του Εράσμους ε, δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν. Πρώτον γιατί ε, είναι πολύ χαμηλή χρηματοδότηση για την κινητικότητα σε αυτό το πλαίσιο και επομένως δεν ε, θα υπάρχουν επαρκή κίνητρα για το δικαστικό σώμα. Το πιο σημαντικό όμως είναι το θέμα της εξοικείωσης των προγραμμάτων αυτών κατάρτισης. Οι δικαστικοί δεν είναι μαθητέ οι οποίοι κάθονται στα φρανία και παρακολουθούν μαθήματα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι όριμοι, επαγγελματίε και έχουν λίγο χρόνο στη διάθεσή του. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο δεν είναι εύκολο να μετακινηθούν αλλά από την άλλη έχουν γνώσεις και θα πρέπει να τους διωθούν ανάλογα κίνητρα ώστε αυτές οι γνώσεις να ε, ε εμπλουτιστούν και με τις νέες γνώσεις που προκύπτουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο και να υπάρχουν ανταλλαγές οι οποίες δεν θα είναι μόνο ανταλλαγές φυκών προσώπων αλλά και ε, διαδικτυακές. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας άλλωστε μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και θα πρέπει να ξεκινάμε και από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι δικαστικοί καθημερινά, τα νέα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν κίνητρο για ε, επαγγελματική εξέλιξη των δικαστικών ώστε να συνεισφέρουν στη συνέχεια ώστε να χρησιμοποιήσουν στη ζωή τους αυτά τα οποία έμαθαν για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ε, της Ευρώπης με θετικό τρόπο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλουμε να προσθέσουμε κάτι νέο ε, τα τμήματα κατάρτιση τα οποία χρησιμοποιούνται μέχρι τούδε και που θεωρούμε ότι δεν επαρκούν για να επιτευχθεί αυτό ο στόχο. Θα θέλαμε να ξέρουμε πόσα κονδύλια διατίθενται, ποια είναι αυτά τα κονδύλια και ε, να εκφράσουμε και κάποιες σε αυτό που αναφέρεται στην ανακοίνωση για μια κεντρική ε, δομή ε, για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού, διότι εμείς είμαστε υπέρ του να έχουμε ένα πρόγραμμα που θα ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω και να μην είναι κεντρικά τα πράγματα θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή νοοτροπία μεταξύ των δικαστικών και των δικηγόρων ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη δικαιοσύνη διότι αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να συνδράμουμε τους ανθρώπους που το ζητούν και δεν θα έχουμε Ευρώπη. Δεν είναι μια χάρτα μόνο για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, είναι μια χάρτα που είναι πάρα πολύ σημαντική για όλο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την τήρηση του χρόνου και για την ιδιαίτερα ενημερωτική εισαγωγή. Παρακαλώ κυρία Γεωργίευα. Thank you, uh, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Κομισιόν. Ευχαριστώ και για την κατάθεση της ερώτησης, για την υποβολή της ερώτησης. Με μεγάλη ευχαρίστηση κάνουμε αυτόν τον διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν προσπαθεί να βελτιώσει την πρόσβαση στην επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών, όχι μόνο για τους δικαστές και τους εισαγγελείς, αλλά για όλους που ασχολούνται με, την νομική, με τα νομικά επαγγέλματα και με συμμετοχή και διαβούλευση των οργανώσεών τους. Τα κράτη-μέλη επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο γιατί έχουν την ευθύνη της επιμόρφωσης των δικαστών κλπ η Κομισιόν αυτή τη στιγμή αποτιμά τι χρηματικά μέσα θα, χρειαζόν, θα χρειάζονταν για να οργανωθεί αυτή η επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών και η ανταλλαγή των γνώσεών τους και θα υποβάλει προτάσεις για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Εν μεταξύ όμως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα μέσα που ήδη διαθέτουμε. Ήδη πήραμε μέτρα για να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η επιμόρφωση των δικαστικών σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι εδώ και πολλά χρόνια οι ενδιαφερόμενοι έχουν ενθαρρυνθεί να αναλαμβάνουν περισσότερα επιμορφωτικά προγράμματα όποτε οργανώνονται διαγωνισμοί, αλλά τα αποτελέσματα μέχρι τώρα ήταν απογοητευτικά η Κομισιόν εκφράζει τη λύπη της ιδιαίτερα γιατί πολύ λίγα ποιοτικά προγράμματα υποβλήθηκαν για την επιμόρφωση των υπαλλήλων δικαστηρίων κλπ. Κλητήρων, δικαστικών κλητήρων και τέτοια. Οι ανταλλαγές των γνώσεων για τα προγράμματα που υπάρχουν στις διάφορες χώρες δεν κατέληξαν φέτος σε κανένα πιλωτικό πρόγραμμα χρειάζονται και άλλες μελέτες για να μας βοηθήσουν να δούμε τι ισχύει για όλα τα νομικά επαγγέλματα και τι αποτελεί ιδιαιτερότητα λαμβάνοντας υπόψη τα οργανωτικά προβλήματα κλάδο αναδικαστικό κλάδο. Για να υπάρξει μια, ένα κοινό δικαστικό κλίμα πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις για να οργανωθούν κοινέ εκδηλώσεις ανάλογα με τα δικαστικά συστήματα της κάθε χώρας το πράγμα το οποίο θα μπορούσε να οργανώσει το μελλοντικό νομικό Ινστιτούτο της Ένωσης. Χρειάζονται βέβαια καλύτερες δομές και έχουν υποβάλει οι δικαστικοί ορισμένα ερωτήματα τα οποία μελετά αυτή τη στιγμή η Κομισιόν όπως τι είδους δραστηριότητες εννοούμε όταν μιλάμε για επιμόρφωση των δικαστικών, τι εργαλεία έχουμε για να κάνουμε την αξιολόγηση, πώς θα δούμε τι προσόντα απαιτούνται και πώς θα γίνει η καλύτερη δυνατή ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών ώστε οι δικαστικοί να μπορούν να επιμορφωθούν και για τα προσόντα που απαιτούνται για να εργαστούν στον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο όπως γλωσσικές γνώσεις ή εργασία σε συνεργασία με τράπεζες και τέτοια ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα συμφέροντα των πολιτών μας. Από τις υπάρχουσες δραστηριότητες δικαστικής επιμόρφωσης θα πάρουμε μαθήματα για να κάνουμε καλύτερη διευθέτηση και νομοθεσία. Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία τα οποία μελετάει η Κομισιόν και που θα αποτελέσουν τη βάση μία ανακοίνωση που θα κάνουμε το 2011 που λέμε. Και θα προβλεφθεί και κατάλληλη χρηματοδότηση βέβαια γιατί έχουμε πολλές ελπίδες για το πρόγραμμα αυτό. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τις συζητήσεις που γίνονται του θέματος και για τη συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κενοβούλιο για αυτό το σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε και τώρα εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων θα αρχίσουμε τον γύρο των δηλώσεων. Πρώτα ο Θαδέος Σιέφκα για δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, <clears throat> η αρχή αμοιβαία αναγνώρισης που είναι θεμελιώδης βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην εμπιστοσύνη στα δικαστικά συστήματα άλλων χωρών. Αυτά όμως θα προκύψουν μόνο από την γνώση των, άλλων, των συστημάτων άλλων ε, χωρών, άλλων δικαιικών και δικαστικών συστημάτων. Η απόκτηση αυτής της γνώσης πρέπει να διευκολυνθεί από μια ειδική πολιτική που θα βασίζεται στην επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών και άλλων προσώπων. Και βέβαια χρειάζεται εξυγχρονισμός και των διδακτικών προγραμμάτων των πανεπιστημίων. Πρέπει να δημιουργηθούν ευρωπαϊκά δίκτυα στα διάφορα δικαστικά συστήματα ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της δικαστικής επιμόρφωσης Σημαντική είναι η προσπάθεια για την ηλεκτρονική επιμόρφωση με κάθε είδους ευφυά συστήματα τα οποία να μπορούν να ε, βοηθούν τους δικαστικούς λειτουργούς να επιλύουν τα νομικά προβλήματα. Με απλές κατευθυντήρες γραμμές για τα δικαστικά συστήματα των χωρών μελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στην σύνταξη και έγκριση των σχετικών κειμένων για την δικαστική επιμόρφωση και κυρίως για πιλωτικά προγράμματα στη βάση των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης. Επίσης σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβουλευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εκπόνηση σχεδίων για τη δημιουργία νέων οργάνων και κυρίως βέβαια της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου. Είναι απαραίτητο, απαραίτητες προσπάθειες αυτές για να, ε, να επιταχυνθεί η επίλυση δικαστικών θεμάτων ε, διαμεθοριακών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι η δεύτερη θητεία μου στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, επομένως κατανοώ πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Το να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο θα είναι αδύνατο χωρίς ε, την επιμόρφωση των νομικών. Και δεν θα πρέπει να λησμονούμε και το ρόλο του δικαστικού σώματος στην προστασία του δικαίου. Οι εθνικοί δικαστές είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποτανθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και πότε υπάρχει παραβίαση σε εθνικό επίπεδο. Οι δικαστές λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Δυστυχώς σήμερα δεν συμβαίνει πάντα κάτι τέτοιο. Επισήμως το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού δικαίου, αλλά ορισμένες περιπτώσεις ε, μας καταδεικνύουν το αντίθετο. Είμαι υπέρ λοιπόν της επιμόρφωσης ε, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δικαστών ή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να υποστηριχθούν ε, καλύτερα από πλευράς χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις δημοσιονομικές προοπτικές για το 2013-2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και που τήρησατε τον χρόνο η κυρία Όλης των Φιλελευθέρων 1,5 λεπτό Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Εμείς οι λίγοι μέλη της Νομικής Επιτροπής μας ε, ενδιαφερόμαστε πολύ για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης αλλά τι νόημα έχει να καθόμαστε εδώ ή στις Βρυξέλλες να ψηφίζουμε καινούριου νόμους εάν οι δικαστές μας δεν γνωρίζουν τους νόμους αυτούς και δεν είναι ικανοί να τους ερμηνεύσουν. Και βέβαια η κατάσταση για την ώρα δεν είναι καλή. Ζητούμε πολλά από τους εθνικούς δικαστές. Θα πρέπει να γνωρίζουν το εθνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αναμένουμε να γνωρίζουν άλλο δαπά δίκαια, δηλαδή των υπολείπων χωρών μελών, να γνωρίζουν γλώσσες, να έχουν γνώση συγκριτικού δικαίου και ούτω καθεξής. Όλα αυτά για να πετύχουν χρειάζονται χρόνο, κόπο, χρήμα. Είναι δύσκολο να επιτευθούν ακόμα και από δικαστές με την καλύτερη θέληση στον κόσμο. Χρειάζονται χρόνο για να τα κάνουν αυτά πράγματα. Προσπαθούμε να κάνουμε κάθε το δυνατόν με διάφορες διασυνδέσεις, προγράμματα, δίκτυα, αλλά και οι χώρες μέλη πρέπει να βοηθήσουν. Εγώ στρέφω τα βλέμματά μου στο μέλλον. Οι νεαροί φοιτητέ δικαίου σήμερα θα είναι οι αυριανοί δικαστέ. Σε αυτούς πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, ώστε οι σπουδέ του να είναι κατάλληλε για να του εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να μπορούν να λειτουργήσουν ω δικαστέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Ακολουθεί ο Γιάννος ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Για να λειτουργεί καλά ο Ευρωπαϊκός Δικαστικός Χώρος πρέπει να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των διαφορετικών νομικών παραδόσεων με αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ δικηγόρων, δικαστών και πολιτών. Οι διαφορές μεταξύ των δικαστικών συστημάτων των χωρών μελών δεν θα έπρεπε να υπονομεύουν τη νομική ασφάλεια των πολιτών ούτε να δυσκολεύουν την ε, άσκηση του δικαιώματός τους σε δίκαια πρόσβαση στις νομικές υπηρεσίες. Γι' αυτό πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης των δικαστικών και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάθε προσπάθεια για να δημιουργήσει ένα δίκτυο νενομισμένων ε, νομικών ιδρυμάτων που να χορηγούν αυτή την εκπαίδευση και επιμόρφωση λαμβάνοντας υπόψη και τον Ευρωπαϊκό Νόμο και τους εθνικούς Κάτι τέτοιο θα βελτίωνε την ποιότητα των νομικών υπηρεσιών στην Ένωση και πρέπει να θεωρηθεί σαν ταπάνη απαραίτητη για να καταλήξουμε σε επίτευξη ενός σημαντικού στόχου, δηλαδή την ικανοποίηση και την ασφάλεια όλων των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. επιτρέψαμε να υπερβείτε λίγο το όριο του χρόνου αγορεύσεως. Ο κύριος Μπαλντάσαρε δεν είναι παρόν. Θα δώσω λόγο στην κυρία Σισίλια Βάικστρομ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Το κοινό μας καθήκον είναι να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη του μέλλοντος που να βασίζεται στις κοινέ μας αξίες και σε μια αμοιβαία εμπιστοσύνη, ο σεβασμό των διαφορών που αποτελεί την ισχύ μας. Οι αξίες αυτές δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο συστάσεων ή απλής νομοθεσίας αλλά πρέπει να βασίζονται σε συνάντηση ανθρώπων ζωντανών. Πρέπει οι άνδρες και οι γυναίκες που ασκούν τις δικαστικές λειτουργίες και τα δικαστικά επαγγέλματα να έχουν τη δυνατότητα να συναντιούνται, να συζητούν, να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Γιατί μόνο με τέτοιες συναντήσεις μπορεί κανείς να καταλάβει τι σημαίνει σεβασμός των διαφορών και μπορεί να πάρει μαθήματα και να κατανοήσει τις διαφορές των συστημάτων. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει περισσότερος διάλογος και περισσότερη αμοιβαία επιμόρφωση και γι' αυτό χρειάζονται ευκαιρίες ανταλλαγών. Ιδιαίτερα δε για τις γυναίκες που είναι η ψυχή του δικαστικού συστήματος στην Ευρώπη. Πρέπει να αναμένουμε πολλά από την Κομισιόν ώστε όλα αυτά να οικοδομήσουν αυτή την Ευρώπη του μέλλοντος που έλεγα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γεωργίευα πάλι. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτά που ακούσαμε εδώ σήμερα συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τις προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε στο μέτρο του δυνατού ένα δίκτυο το οποίο θα επιτρέψει τους επαγγελματίες να μάθουν από τις δεξιότητες και τις δυνατότητες των καλύτερων αλλά και να αποτελέσει και μια πλατφόρμα για να έχουμε επιμόρφωση σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να έχουμε ένα ενεργό δίκτυο όπως για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δικαστών, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο Κατάρτισης, ε, την Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και ούτω καθεξής. Έγινε μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Ακούσαμε ότι πρέπει να εστιάσουμε στο μέλλον και αυτό φυσικά είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ερώτημα είναι πώς θα το εφαρμόσει. πώς θα εξελιχθούν τα προγράμματα κατάρτισης το 2011, αλλά και με την ανακοίνωση για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προεπτικές. Θα ήθελα να κάνω μια πολύ συγκεκριμένη παρατήρηση. Με χαρά μου ενημερώνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα ξεκινήσει μια δικτυακή πύλη για το e-Justice στις 16 Ιουλίου, διότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε τη νέα ανακοίνωση. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή. Άλλωστε, μας ενδιαφέρει η καλύτερη εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά θα πρέπει να αυξηθεί και η εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό δίκτυο, ώστε να βασίζονται στη συλλογική πρόοδο, η οποία έχει ως τελικό αποδέκτη τους πολίτες μας. Θα σταματήσω εδώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που βρίσκεστε εδώ στο Προεδρείο. Νομίζω ότι ε, τα πήγατε πολύ καλά. Ξεκινήσαμε στις 9 και 5 και φαίνεται ότι θα τελειώσουμε 12 παρα 5. 5 λεπτά λοιπόν πριν <laughs> από τη λήξη της συνεδρίασης. Να σας συγχαρώ λοιπόν και ελπίζω στο μέλλον να είστε τόσο οργανωτικός όσο ήσασταν και σήμερα. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Εύχομαι και εγώ η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου